και θα συνεργαστούμε στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για τι μελλοντικέ προτάσει οι οποίες όπως είπα θα κατευθούν τον Οκτώβριο. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση αύριο στις 11.30 ψηφοφορία. Στην ημερήσια διάταξη τώρα έχουμε την έκθεση της κυρίας Γιανακουδάκη για τις γυναίκες της ηθήνουσες θέσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια λοιπόν για τέσσερα λεπτά. Παρακαλώ. Thank you. As governments face economic... Με την οικονομική αναταραχή που αντιμετωπίζουν οι κυβερνήσεις είναι σημαντικό να αξιοποιήσουμε τους πόρους που έχουμε με τον καλύτερο τρόπο. Οι εταιρείε και οι επιχειρήσει είναι ένα τέτοιο πόρο που δημιουργούν πλούτο που χρειάζεται σε μια σφίζουσα επιτυχημένη οικονομία. Ε, σήμερα εξετάζουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βλέπουμε ότι δικούνται κυρίως από τους άνδρες. Αυτό σημαίνει ότι ένα κομμάτι του πληθυσμού δεν αξιοποιεί το δυναμικό. Ε, η έκθεση αυτή αναφέρεται στη θέση των γυναικών στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δέχεται τα προβλήματα και αναγνωρίζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην επιτέψη των στόχων τους. Επίσης η έκθεση αναγνωρίζει τη συμβολή των γυναικών στην απασχόληση. Ε, τόσο στην τοπική κοινότητα όσο και στην ε, ευρωπαϊκή οικονομία και καταδεικνύει ότι οι γυναίκες έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν το ρόλο που θα παίξουν είτε στο σπίτι είτε στην κοινότητα όπου ζουν. Πολλές γυναίκες ε, θα πρέπει να κάνουν ακροβασίες για να επιτύχουν ε, παράλληλα με τις υποχρεώσεις στην οικογένεια. Ο στόχος της οικογένειας, της έκθεσης είναι να θεσπίσει πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις που θα μπορούσαν να υιοθετήσουν αν το επιθυμούν τα κράτη-μέλη για να βοηθήσουν τις γυναίκες. Βεβαίως υπάρχει διαφορετική προσέγγιση προς τη στις γυναίκες που έχουν επιχειρήσεις. Ε, υπάρχει διαφορά στην υποστήριξη που δίνουν τα κράτη-μέλη. Ε, καθώς έκανα την έρευνά μου είδα ότι υπάρχουν δυσκολίες ε, για να στήσουν μια επιχείρηση οι γυναίκες. Παρόμοια στα κράτη-μέλη. Πολλές φορές δεν γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν για να στήσουν μια επιχείρηση. Δεν έχουν την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους ή δεν ξέρουν πού θα πρέπει να απευθυνθούν. Και τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα δεν τις στηρίζουν συχνά. Ε, έκανα, προτείνω λοιπόν κάποιε τροπολογίε ε, όπω ε, καλύτερη χρήση των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων που υπάρχουν για τι γυναίκε επιχειρηματίε, ούτω ώστε να υπάρχει δίκαιη και ισότιμη πρόσβαση στην οικονομική υποστήριξη. Επίση, οι νέε επιχειρηματίε θα πρέπει να εκπαιδεύονται καλύτερα, θα πρέπει να ενθαρρύνονται προγράμματα σε πανεπιστήμια τα οποία θα απευθύνονται σε νέε επιχειρηματίε. Θα πρέπει επίσης να υπογραμμίσουμε τη γυναίκα την σημασία εργασία των γυναικών πρεσβυρών γιατί ε, εμπνέουν, αποτελούν πηγή έμπνευση για τις νέες γυναίκες να δημιουργήσουν επιχειρήσεις. Ε, καταρτίζοντας την έκθεση, κατά την κατάρτιση θέλω να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές διότι νομίζω ότι ενίσχυσαν την έκθεση με τη συμβολή τους θα γίνουν χωριστές ψηφοφορίε ε, στις παραγράφους 44 ε, και 46, 34, 46 και 46 για τους ε, Ρώμ, τι μετανάστριε και την ισόρροπη εκπροσώπηση στα συμβούλια, διοικητικά συμβούλια. Όλα αυτά τα θέματα είναι πολύ σημαντικά, αυτό δικαίω, Αλλά δεν είναι τόσο σημαντικά σε μια έκθεση που ε, ε, εστιάζει στις γυναίκες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν δεν θα υποστηρίξω αυτές τις ε, χωριστές ψηφοφορίες. Ως γυναίκα που επί 25 χρόνια είχα τη δική μου επιχείρηση, γνωρίζω από πρώτο χέρι τα προβλήματα που μπορούν να αντιμετωπίσουν οι γυναίκες όταν προσπαθούν να δημιουργήσουν μια βιώσιμη μικρομεσαία επιχείρηση. Ελπίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει την έκθεση και τα κράτη-μέλη ελπίζω να χρησιμοποιήσουν την έκθεση έκθεση ως βάση για να υποστηρίξουν γυναίκες που θέλουν να ε, εξελιχθούν σε αυτό το τομέα. Γιατί παρά όλες τις, ε, τους, όλους τους περιορισμούς, ε, οι γυναίκες απέδειξαν ότι είναι πάνω πιο πολύ από ικανές όταν λειτουργούν ως επιχειρηματίες. Θα πρέπει λοιπόν και μια έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από άλλα μέσα να τις υποστηρίξουμε. Δεν θα ενθαρρυνθούν μόνο έτσι να περάσουν στον κόσμο των επιχειρήσεων, αλλά θα βεβαιωθούμε όταν θα κάνουν το βήμα θα υπάρχουν ίσοι κανόνες του ε, παιχνιδιού και δεν θα γίνονται διακρίσεις μεταξύ φίλων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μπάστος. Ευχαριστώ κύριε κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς να συγχαρώ την εισηγήτρια για την εξαιρετική της δουλειά και θα ήθελα να την ευχαριστήσω και γιατί ήταν ιδιαίτερα ανοιχτή και επέδειξε πνεύμα συνεργασίας κατά την κατάθεση τροπολογιών οι οποίες έτυχαν και ευρεία συνένεσης. Το να μιλούμε σήμερα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρηματικότητα, είτε είναι των ανδρών είτε των γυναικών, είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη δεδομένων των μεγάλων δυσκολιών που αντιμετώπισαν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια. Εξακολουθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να είναι σημαντική πηγή δημιουργία θέσεων εργασία και δυνατότητα ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα λοιπόν για τι γυναίκε επιχειρηματίε, διότι υπάρχουν τεράστιε δυνατότητε, ένα τεράστιο δυναμικό που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε και αυτό φυσικά μπορεί να βοηθήσει και την απασχόληση. Η εισηγήτρια ζητά να δοθούν και κίνητρα ώστε να μπορέσουν οι γυναίκες να συμφιλιώσουν οικογενειακό και επαγγελματικό βίο, δημιουργώντας έτσι καλύτερες επιχειρήσεις για τις γυναίκες. Ε, χαιρόμαστε ιδιαίτερα και για τις συστάσεις για τον τρόπο χρηματοδότησης και των ε, χρηματοοικονομικών μέσων που υπάρχουν στη διάθεσή τους και όπως για παράδειγμα τη δυνατότητα μικροπιστώσεων. Εδώ θα πρέπει να επαναλάβουμε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Progress, το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει. Θα ήθελα επίσης να σταθώ λίγο και στο περιεχόμενο της παραγράφου 46. Για νομικούς λόγους και λόγους συνέπειας θα ψηφίσουμε χωριστά τη συγκεκριμένη παράγραφο. Δεν είμαστε αντίθετοι σε καμία περίπτωση στην ισορροπημένη συμμετοχή γυναικών και νέων στα ε, διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων. Δεν είναι αυτό το νόημα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους τους αδέλφους ότι προβλέπεται ένα λεπτό ομιλίας για τη διαδικασια κατς ΚΑΤΣ-ΔΙΑΕ. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας ζητήσω να τηρείτε ε, τα χρονοδιαγράμματα. Ο κύριος Νικολα... Μικολάσικ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η ανεξάρτητη απασχόληση είναι ευέλικτη σε σύγκριση με ε, ένα κλασικό επάγγελμα και έτσι η ανεξαρτησία αυτή επιτρέπει το συγκερασμό οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Η οικογένεια είναι βέβαια η βάση της κοινωνίας. Είναι λυπηρό που μία στις δέκα γυναίκες στην Ευρώπη είναι επιχειρηματίας παρόλο που οι γυναίκες είναι το 60% των αποφύτων του Πανεπιστημίου. Τα κράτη-μέλη λοιπόν, αλλά και οι επιμέρους ε, δημόσιες υπηρεσίες ε, πρέπει να βελτιώσουν τις προϋποθέσεις που θέτουν για τις γυναίκες όπως ε, ειδικέ επιδοτήσεις για γυναίκες, μικροπιστώσεις σε γυναίκες που θέλουν να ιδρύσουν τη μικρή τους επιχείρηση και παρόμοια μέτρα εδώ πρέπει να απευθύνουμε έκκληση στα κράτη-μέλη, ώστε με τη σειρά τους να ασκήσουν πιέσεις προς τις τράπεζες ε, για τέτοιου είδους μέτρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Παντσίλα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η τρέχουσα χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση η οποία πλήττει την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιτείνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηματίες, ιδιαίτερα στα πρώιμα στάδια της επιχείρησής τους. Γνωρίζουμε όλοι πόσο σημαντικές είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την ευρωπαϊκή οικονομία διότι άνω το 25% των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, δημιουργούνται από άνεργους ανθρώπους. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει στο μελλοντικό προϋπολογισμό της Ένωσης ε, υποστήριξη για γυναίκες επιχειρηματίες και θα πρέπει να δίνεται χωρίς καμία διάκριση η χρηματοδότηση οι πρωτοβουλίες για τις γυναίκες θα πρέπει να προάγονται περισσότερο στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, ιδίως όταν πρόκειται για ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Φλασίκοβα μπαίνω. Κυρία, κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, Δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι και σήμερα εξακολουθούν οι διακρίσεις σε βάρος των γυναικών στην αγορά εργασίας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός. Ε, είναι πολύ πιο δύσκολο μια γυναίκα να ιδρύσει μια μικρομεσαία επιχείρηση. Ε, υπάρχουν πολλά εμπόδια και ίσως ό,τι αφορά την πρόσβαση στην ενημέρωση πληροφόρηση και γι' αυτό οι δυνατότητες των γυναικών περιορίζονται πολύ. Και σε αυτόν τον τομέα. Οι ικανότητες των γυναικών αποτελούν πολύτιμο ε, δυναμικό για ολόκληρη την κοινωνία. Πρέπει να δώσουμε κίνητρα στις γυναίκες να δραστηριοποιηθούν ως επιχειρηματίες, θα πρέπει να λάβουμε μέτρα για ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών εδώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Τικάου. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι λόγω της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης οι γυναίκες επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρότερα προβλήματα. Καλούμε την Κομισιόν, τα κράτη-μέλη και τις ε, τοπικές αρχές λοιπόν να αξιοποιήσουν τις χρηματοδοτικές δυνατότητες που υπάρχουν όπως ε, το μέσο Progress το οποίο παρέχει 25.000 ευρώ σε πολύ μικρές επιχειρήσεις. Για να γίνουν επιχειρηματίες οι γυναίκες θα πρέπει να τους επιτραπεί η πρόσβαση στην τεχνολογία της πληροφορίας, της επικοινωνίας. Είναι σημαντικό οι δραστήριες ενεργές γυναίκες να έχουν και υπηρεσίες φύλαξης παιδιών. Καλό την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη να δώσουν έμφαση και στις γυναίκες άνω των 50 και να βοηθήσουν και εκείνες να δραστηριοποιηθούν λαμβάνοντας υπόψη προγράμματα τα οποία απευθύνονται σε αυτή την κατηγορία των γυναικών. Ευχαριστώ. Κυρία Φιγκερέιδο. Ευχαριστώ πολύ. Η τωρινή κρίση ίσως ε, πλήττει περισσότερο τις γυναίκες, ιδιαίτερα τις γυναίκες χαμηλών εισοδημάτων. Το χαμηλό επίπεδο της απασχόλησης και η ψηλή επισφάλεια των χαμηλών, χαμηλά αμοιβωμένων ε, επαγγελμάτων δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη όξυνση της εκμετάλλευσης και των διακρίσεων. Πάνω σε αυτή τη βάση πολλές γυναίκες ε, μπαίνουν στον πειρασμό να κάνουν ψεύδο απασχόληση. Περνούν δηλαδή σε ένα ψεύδο επιχειρηματικό κλάδο. Ε, πράγμα που σημαίνει ότι δουλεύουν περισσότερο ενώ ε, οι εργοδότες ε, απαλλάσσονται από τις κοινωνικές υποχρεώσεις που θα είχαν. Αυτό πρέπει να καταπολεμηθεί. Όντως υπάρχουν γυναίκες σε μικρές επιχειρήσεις, σε πολύ μικρές επιχειρήσεις που χρήζουν υποστήριξης και θα πρέπει να τις υπερασπιστούμε απέναντι σε κάθε μορφή ε, διακρίσεων. Ε, άρα λοιπόν πράγματι και εγώ προσυπογράφω ε, ορισμένα από τα μέτρα που αναφέρονται εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Μπασέσκου. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στην ανάπτυξη. Δυστυχώς υπάρχει ακόμα ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Οι γυναίκες είναι μόνο το 30% των Ευρωπαίων επιχειρηματιών. Πρόκειται για μια διάκριση η οποία είναι εις βάρος και των γυναικών αλλά και της οικονομίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται όλο ένα και περισσότερα προγράμματα τα οποία να δώσουν κίνητρα και να υποστηρίξουν τις γυναίκες επιχειρηματίες. Γι' αυτό υποστηρίζω τη δημιουργία ενός οργανισμού ο οποίος θα υποστηρίζει τις επιχειρήσεις που ε, διαχειρίζονται γυναίκες. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε μιας μορφής ρεάλ πολιτική για τις γυναίκες επιχειρηματίες. Οι γυναίκες επιχειρηματίες είναι ένας πόρος ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιείται πολύ πιο αποδοτικά σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πάσκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, εκτιμώ ιδιαίτερα το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταβάλει προσπάθειες για τη βελτίωση της θέσης της γυναικός στην κοινωνία. Σε διάφορες εκθέσει και συστάσει. προτρέπουμε τις χώρες μέλη να θεσπίσουν καλύτερα νομοθετικά μέτρα για, υπέρ των γυναικών για να μπορούν αυτές να επιτύχουν περισσότερα και στη δημόσια διοίκηση και στον επιχειρηματικό τομέα αλλά και στην οικογενειακή ζωή. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι αποδίδουν οι προσπάθειες αυτές του Ευρωκοινοβουλίου. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τις γυναίκες ως επιχειρηματίες, θα πρέπει να μπορούμε να αξιολογήσουμε καλύτερα και το λεγόμενο feedback. Να δούμε δηλαδή ποια από τα μέτρα που ζητούμε είναι επιτυχέστερα και πια αποτυγχάνουν. Μετά από μια τέτοια αξιολόγηση θα μπορέσουμε να προτείνουμε καλύτερα μέτρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τσάρος. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση δημιούργησε τεράστια προβλήματα στους πληθυσμούς μας. Ιδιαίτερα οι γυναίκες κάτω των 50 ετών πλήττονται. Υπάρχουν επιχειρηματίες, υπάρχουν ε, ως ποσοστό αρκετές γυναίκες που δραστηριοποιούνται σε μικρές και πολύμνες επιχειρήσεις αλλά ε, χρειάζεται περισσότερη υποστήριξη για να συνεχίσουν οι γυναίκες αυτές την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Γι' αυτό χρειάζονται ενωσιακά κονδύλια και χρειάζεται αυτά να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο. Ειδικότερα πρέπει να βοηθηθούν οι γυναίκες ε, ώστε να μπορέσουν να συμβιβάσουν την οικογένεια με το επάγγελμα. Επίσης ε, θα πρέπει να ε, υποστηριχθούν να βελτιώσουν τις ικανότητές τους. Είναι σημαντικό το έργο αυτό των γυναικών να εκτιμηθεί όπως πρέπει και να βρουν μια, τη θέση που τους ε, ανήκει στην αγορά εργασίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό ε, εν ώψη της κρίσης που συνεχίζεται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Νεβιτάλοβα. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Οι γυναίκες δυσκολεύονται πολύ στην αγορά εργασίας ε, γιατί οι διακρίσεις εξακολουθούν να υφίστανται λόγω φύλου, ε, δυσκολιών από την οικογένεια κλπ. Πολλές γυναίκες δεν έχουν το θάρρος, την τόλμη να ε, γίνουν επιχειρηματίες. Χαιρετίζω λοιπόν γι' αυτό το λόγο την έκθεση γιατί είναι αναγκαίο να δοθούν κίνητρα στις γυναίκες να ξέρουν ότι θα έχουν την υποστήριξή μας ε, χαιρετίζω την πρωτοβουλία στα πλαίσια του προγράμματος Εράσμους την ε, εκπαίδευση των νέων επιχειρηματιών γυναικών. Απευθύνω έκκληση στα κράτη-μέλη μας ώστε να βρουν πόρους για να προωθήσουν τις γυναίκες περισσότερο και να έχουν ίδιες ευκαιρίες και ίδια πρόσβαση στα ε, οικονομικά, στους οικονομικούς πόρους. Καλό, είναι να γίνει κάτι και για την, ε, στις συμβουλευτικές υπηρεσίες οι πλατφόρμες σε διεθνές επίπεδο χρειάζονται για να λύνονται τα πρακτικά προβλήματα των γυναικών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Παπαδοπούλου. Σωστά η Ευρωπαϊκή. Ευχαριστώ. Τη γυναικεία επιχειρηματικότητα συγχρηματοδοτώντα με μικροπιστώσει καινοτόμε μικρομεσαίε επιχειρήσει. Ωστόσο, είναι η ώρα να ανεβάσει ταχύτητα πέραν από την ανάγκη καταπολέμησης έφυλων ανισοτήτων και συμφιλίωση οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων έμφαση πρέπει να δοθεί στην οικονομική και εκπαιδευτική στήριξη των γυναικών επιχειρηματιών με προγράμματα επιχειρηματική καθοδήγησης στην αφετηρία αλλά και στη διάρκεια των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων εξοικείωση με τι νέε τεχνολογίε των πληροφοριών και επικοινωνιών γιατί ανοίγουν νέου ορίζοντε και ευκαιρίε στην καινοτόμα απασχόληση και τέλο συμπερίληψη ειδικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων σε σχολικά και πανεπιστημιακά προγράμματα και ανάδειξη θετικών προτύπων για τόνωση τη αυτοπεποίθηση και ανάπτυξη τη επιχειρηματική δραστηριότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ για τη σημαντική αυτή έκθεση. Εξακολουθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να επιχειρούν περισσότεροι άνδρες από γυναίκες. Θα ήταν λοιπόν σημαντικό να δημιουργηθεί ένα παρόμοιο με το αμερικανικό ε, γραφείο για την ε, γυναική επιχειρηματικότητα. Οι γυναίκες μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα και μάλιστα ταυτόχρονα. Είναι πολύ σημαντικό για τις σημερινές κοινωνίες περισσότερες γυναίκες να μπουν στον επιχειρηματικό κόσμο με προώθησή τους και στο τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ευχαριστώ. Grazie. La parola al ο Επίτροπος Ταγιάννη τώρα, παρακαλώ. Έχουμε προτείνει συγκεκριμένες δράσεις για την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του Small Business Act για την Ευρώπη. Η πρώτη δράση ήταν η δημιουργία ενός δικτύου των πρεσβυρών της γυναικείας επιχειρηματικότητας το 2009. Ζητήσαμε επίσης από τους επιχειρηματίες να κάνουν επιτόπου εκστρατείες για να παρακινήσουν τις γυναίκες όλων των ηλικιών να αναλάβουν επιχειρηματική δράση. Αυτά είναι πολύ σημαντικά, να έχουν πρότυπα δηλαδή οι γυναίκες για να ξεκινήσουν μια νέα επιχείρηση. Σήμερα έχουμε 320 πρέσβυρες σε 22 ευρωπαϊκές χώρες. Το δίκτυο αυτό λοιπόν υπήρξε επιτυχία από την πρώτη του χρονιά ξεπέρασε τους στόχους του δημιουργώντας πολλές γυναικές επιχειρήσεις σε πολλές ε, ε, χώρες. Οι πρέσβυρες αυτές μάλιστα ξεπέρασαν και τα καθήκοντά τους κάνοντας εκστρατείες υπέρ της γυναικής επιχειρηματικότητας. Συμμετέσχουν ενεργά για την προώθηση των νέων επιχειρήσεων. Χάρη στην δουλειά τους στις έξι χώρες που συμμετέχουν γιατί δεν έχουμε δεδομένα για άλλες χώρες, πάνω από 110 νέες επιχειρήσεις που διευθύνονται από γυναίκες έχουν ήδη δημιουργηθεί. Η Κομισιόν για τις 15 Νοεμβρίου προωθεί το ξεκίνημα του έτους της γυναίκας επιχειρηματίου. Θα κινητοποιήσουμε τις γυναίκες επιχειρηματίες για να δράσουν έτσι ώστε να προσελκύσουν και άλλες γυναίκες επιχειρηματίες προσφέροντάς τους συμβουλές για το λεγόμενο start-up, για το ξεκίνημα δηλαδή και την πρόθεση της επιχειρήσεώς τους. Θα επιλεγούν στο εθνικό επίπεδο από τα συμμετέχοντα μέλη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Ψηφοφορία αύριο στις 11.30. Και τώρα στην ημερήσια διάταξη έχουμε την έκθεση της Edith Bauer για την κατάσταση των γυναικών που πλησιάζουν την ηλικία συνταξιοδότησης.